Domnul președinte. Stimați colegi, ședința... Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την πρώτη έκθεση που προβλέπετε σήμερα το απόγευμα. Θα σας ενημερώσω ότι είναι στη διάθεσή σας τα πρακτικά και τα κείμενα που υιοθετήθηκαν εχθές. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι.